Okay, friends. Uh, we Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αρχίζει το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Έχουμε ψηφοφορίες. Έγκριση γνωμοδότησης υπομορφή επιστολή σχετικά με τις αιτήσει κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Είναι και ονομαστική λοιπόν η κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο σημείο 11 για την επιστολή σχετικά με το Ταμείο Καταπολέμησης τη αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Πέρασε. Εγκρίνεται 34-2. Συνεχίζουμε. Έγκριση ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη του κυρίου Χέντελ. Σας δίνω ένα λεπτό να λάβετε τις θέσεις σας και να βάλετε τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Now we'll start uh, uh, with the, the European Solidarity Corps. Έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ψηφίζουμε τροπολογία παριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται έλεγχο θέλετε παρακαλώ. The Solidarity Corps. E oh, sorry. sorry. Uh, EPP is one many. Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται με 23 ψήφους. Η τροπολογία παριθμό 2 έχει καταπέσει διότι εγκρίθηκε η παρθμονένα και η 3 επίσης. 4 και 5 επίσης, όλα αυτά έχουν καταπέσει και πάμε στην τροπολογία παρθμών 6. Ψηφί περ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά στην ελέγξουμε και αυτή. Uh, Εγκρίνεται 24 υπέρ 18 κατά. Έξι διαφορά. Ε, Θέλουμε, λέει η κυρία Στάινρουκ, να αποσύρουμε την τροπολογία μας υπαριθμών 7, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και πρέπει να εγερθούμε γι' αυτό. Uh, λοιπόν, αποσύρεται η τροπολογία 7 εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και η επόμενη τροπολογία επίσης. Να σας εξηγήσω από πλευρά των Πρασίνων ότι θέλουμε να αποσύρουμε ε, την τροπολογία υπαριθμών 8. Κάπου σε κάποια λίστα ψηφοφορίας λέει 9, ναι, αλλά είναι 8 των πρασίνων τροπολογία, λέει η κυρία Λάμπερτ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε πλέον την τροπολογία 9 μόνο ε, να ψηφίσουμε. You maintain that. Uh, okay. We vote Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεν απεσύρθη αυτή η τροπολογία. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 39 ψήφους. Η τροπολογία 11 καταπίπτει. Η 10 προηγουμένως όμως. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψήφι κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Προχωρούμε. Microphone. 11, those in favor. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Η 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 14. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 υπέρ. Φόλς λέει εδώ, καταπίπτει. Amendment 16. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήταν σαφές, αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε, σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 36 ψήφους. Η τροπολογία 17 καταπίπτει, όπως και 18. Ψηφίζουμε τη 18. Αρχίζει ψηφοφορία. And uh, the vote is now closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 26 ψήφοι κατά. Η τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. 42 υπέρ. Η τροπολογία 20 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 υπέρ αυτή κάναμε τώρα. Α, συγγνώμη. Ε, ψηφίζουμε το σύνολο τώρα, όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. yeah. very quickly. Πάρα πολύ γρήγορα. Η τροπολογία 19 λέει πως υπάρχει πρόθεση να αποφευχτεί ο δόλος και η απάτη. Duplicity λέει στα αγγλικά. Υποθέτω ότι εννοείται duplication που είναι οι επικαλύψεις και οι διπλές δουλειές. Ναι, ωραία, είναι μια γλωσσική διόρθωση αυτή. Θα το δουν οι αρμόδιοι για να διαγράψουν την επίμαχη λέξη. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. proceed with our uh, collaborative Yes, we shall proceed with the... Uh, λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η συνεργατική οικονομία. Αρχίζουμε από το συμβιβασμό 4. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία Συμβιβαστική πάντα 6 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 Θέλετε έλεγχο για την 11. Παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι. Συμβαστική 2 ψήφοι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για τη 14. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Λίγη. And it's carried by 26 votes. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 τώρα ψήφιπε κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 22 ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 22 ψήφιπε κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 κατά τμήματα τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι έχει απορριφθεί αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονική απαρίθευση για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας παριθμών 26. Αρχίζει η ψηφοφορία και λίγη τώρα. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 27 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχει 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθών 36 υπέρ. Α, όχι το πρώτο τμήμα, διότι έχει και τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα υπέρ, κατά, αποχές Μάλλον έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγ... απορρίπτεται. Η συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 103. Έχουμε μια προφορική τροπολογία εδώ υπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 109 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 109. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Η 110 τροπολογία ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 36 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ όχι, διορθώνει η Πρόεδρο, συγγνώμη. Πέρασα μια τροπολογία. 133 επέ, 133, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είμαστε σε 134 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνές, ωραία. Ε, ελέγχουμε την 134 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο. Διαφορά. Η τροπολογία 135 ψήφι πέ, κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Θέλετε έλεγχο. Για ποια τροπολογία, την 136. Έχει καταπέσει. 135. I can't hear. Is it 135 you want to check? Okay, we check. Α, την 135 θέλετε να ελέγξουμε. Μάλιστα. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Yeah. Mm -hmm εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. ψήφι πέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Συμβαστική επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ήρθε η ώρα της τελικής ψηφοφορίας ονομαστικά για το σύνολο του σχεδίου όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ, μία κατά και 8 αποχές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, κύριε Σούστερ. Uh, We don't have it in colors now. You have it in color for you. Is it same now? Ah.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 Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός παρελθόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ο συμβιβασμός 2. Τροπολογία 37, σελίδα 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μαζί ψηφίσουμε τη 40 και 41. 4 και 40, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και 47 μαζί υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται, αλλά το ελέγχουμε. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά Τις τροπολογίες 7 και 47. Τις ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά μαζί. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Με τέσσερις ψήφους παραπάνω. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 Όχι, ψηφίζουμε την 57 και 59 μαζί. Διορθώνει πρόεδρος υπέρ κατά, εποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 9 και 10 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 56 και 58 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτονται. Τροπολογία 60. Ας τσεκάρουμε όμως ηλεκτρονικά την ε, τροπολογία 11. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτονται με δύο ψήφους παραπάνω. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 13 ηλεκτρονικά ψηφίσουμε τώρα πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η καταπίπτει 61. Πάμε στην 62. Τσεκάρουμε φωνικά τη 14. τη φοφορία, Εγκρίνεται με μια ψήφο παραπάνω. ή 61 καταπίπτει γιατί είναι διορθωτική. Ήταν λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών. Πάμε στην τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με την 62, την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 16 και 17 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογίες. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 69 ψηφίσουμε και αυτήν 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και μετά. Πάμε στην αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 18 υπέρ Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. Τον κύριο Καλβέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε τώρα. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε για την καλή και αποτελεσματική προσπάθεια που κάνετε, κύριε Και τώρα Περιμένω τον επόμενο κατάλογο. Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Συμβαστική S, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, η Ει-Ειτς υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική G, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G εγκρίνεται. I εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι Απορρίπτεται, αλλά στην με ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με πέντε ψήφους συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 προφορική υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και U. 78 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται αλλά μπορούμε να την ε, τσεκάρουμε ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται κατά τέσσερις ψήφους Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z εγκρίνεται Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές. Για να την τσεκάρουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική AA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Στο σχέδιο γνωμοδότησης άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο. Για την εισηγήτρια, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. And those of you who are not running, uh, we'll proceed with, uh, Θα προχωρήσουμε. Με το σημείο 17 δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Θα περιμένω ένα λεπτό να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα. Okay, friends. Uh, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, to to next... Αν δεν θέλετε να ακούσετε το επόμενο θέμα στην μερίσια διάταξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης, so παρακαλείστε να αποχωρήσετε ησύχως για να ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Λαβριέ. sorry, friends, but... Κοιτάξτε, πρέπει να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και την ευκαιρία να ακούγεται η φωνή του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης και είχα την ευκαιρία να σας το παρουσιάσω στις 28 Φεβρουαρίου συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, πρόκειται για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και ένα σχέδιο κανονισμού του λεγόμενου Omnibus. Η Επιτροπή μας έχει την αρμοδιότητα για τέσσερα άρθρα, για τέσσερις δημοσιονομικούς κανονισμούς. Το 263 θυμίζω αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την καινοτομία, την κοινωνική. Το άρθρο 266 που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ESF, το 271 που αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το άρθρο 273 που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, βοήθεια στους πλέον απόρους. Τα υπόλοιπα άρθρα δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας, οπότε εξετάζονται σε άλλες καθήλυνα αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το σχέδιο λοιπόν γνωμοδότησης που σας προτείνω σέβεται και εμβαθύνει τους άξονες της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απλούστευση που θέλησα να τη συνδέσω με πιο μεγάλη ε, αποτελεσματικότητα στη χρήση των ε, οικονομικών πόρων. Σήμερα είναι πάρα πολύ περίπλοκοι οι κανόνες, οι δημοσιονομικοί και είναι δύσκολο να εκτελούνται τα προγράμματα. Είναι δύσκολο και για τους διαχειριστές και για τους δικαιούχους που τελικά είναι μικρομεσαίοι και ε, οι πολίτες. Στις εκθέσεις ε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ε, ζητεί ευρύτερη χρήση ε, των ε, διαφόρων εκδοχών για το απλοποιημένο κόστος. Έτσι θα μειώνονται και τα σφάλματα που κάνουν οι διαχειριστές και θα βελτιωθεί γενικότερα η αποτελεσματικότητα της χρήσης και της πρόσβασης στους πόρους αυτούς. Αυτή λοιπόν η διευκόλυνση, η γνώση και η χρήση των ταμείων είναι σημαντικό πολιτικό διακύβευμα γιατί έτσι δείχνει ότι είναι πιο αποτελεσματική η Ένωση στα μάτια των κρατών μελών, των επιχειρήσεων και κυρίως των πολιτών. Οι τροπολογίε στο σχέδιο γνωμοδότησή μου είναι ε, προ την ίδια κατεύθυνση για το άρθρο 263. Οι τροπολογίε μου είναι κυρίω υπέρ μια καλύτερη και μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των πόρων του Ταμείου για την Καινοτομία. Δηλαδή, αν δεν απορροφούνται σε ένα χρόνο νη, ε, σε ένα οικονομικό έτος νη δηλαδή, να μπορούν να μεταφέρονται οι πιστώσεις στον επόμενο χρόνο νη συνένα για να μπορεί να ενισχύεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επίσης, ο κανονισμός αυτός, μάλλον ο προϋπολογισμός, δεν θα έχει αυστηρή κατανομή μεταξύ των τριών κλάδων, αλλά ένα ελάχιστο κατόφλι. Για το 266, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θέλω να γενικεύσω ε, τις ε, επιλογές και τις εκδοχές απλουστευμένου κόστους για να υπάρχει λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος και να μειωθούν και τα σφάλματα. Επίσης, Ζητάω να υπάρξει μια οροφή, ένα πλαφόν 150.000 ευρώ για τις ενισχύσεις, ενώ είναι 50.000 το προτινόμενο σήμερα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να γίνει 100.000. Επίσης ζητώ παρέκκληση για τις κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ε, σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις και βαριές. De minimis λέγεται αυτή η εξαίρεση, η παρέκκληση και θα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει όπως αποφασίζει για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ορισμένων περιφερειών μας όπως θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, την περιφέρεια Eau de France, που είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Από το άρθρο 271, Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Οι προτάσεις μου και οι τροπολογίες μου προβλέπουν τη δυνατότητα, τα κράτη-μέλη, να έχουν δυνατότητα να αποβάλουν αίτηση για σύνολο επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο ή στην ίδια περιοχή. Δηλαδή θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται και μικρομεσαίες εκεί. Επίση, ζητώ να είναι η απόκριση 7 μέρε το πολύ μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το άρθρο 273 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας στους Απόρους ε, οι τροπολογίε μου προς την ίδια κατεύθυνση ζητούν ε, πλαφόν 150.000 ευρώ. Επίσης, ε, τροποποιώ το 265, κάνω τροπολογίες δηλαδή που δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Θέλησα να ζητήσω την ίδια οροφή για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία στρατηγικών επενδύσεων. Έτσι, γενικότερα, έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα που αναθεωρούμε τις ε, πολιτικές και τους προσανατολισμούς. Είναι πολλές υποχρεώσεις, πολλή η λογιστική και πολλές φορές αποκομμένοι από ορισμένες ε, περιφερειακές πραγματικότητες. Χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική επενδύσεων, μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη απλούστευση ε, και στην ε, κατανομή των πόρων αλλά και στη συνδιαχείριση. Γενικά ε, αυτό είναι το πνεύμα του σχεδίου γνωμοδότησής μου. Ε, θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας και περιμένω και τις τροπολογίες σας. Αν δεν απατώμε μέχρι τις 28 Μαρτίου έχουμε προθεσμία κατάθεσης έτσι ώστε από κοινού να μπορέσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus. Σας ευχαριστώ για την τόσο μεγάλη προσοχή και για την τόση πολυάριθμη παρουσία. Παραλίγο να πω ότι καλύτερη είναι εδώ, αλλά κρατήθηκα. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις. Εστιάζει στα βασικά θέματα που είναι προβληματικά στην πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες και, και για την αρχική πρόταση Και θα έχουμε να προτείνουμε στον εισηγητή διάφορε δικέ μα τροπολογίε. Καταρχά, Πρόεδρε, η γενική παρουσίαση της πρότασης υποτίθεται ότι προωθεί την ε, απλούστευση και την ευελιξία. Άρα είναι τεχνικής φύσεως. Ε, με αυτό όμω εμεί διαφωνούμε κάθετα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση Αντίθετα, είναι πολύ πολιτική, πολύ πολιτικοποιημένη, γιατί συμπεριλαμβάνει μίσονες αλλαγές για τον συνδυασμό των ταμείων και την μεταφορά των κονδυλίων των ταμείων. Είναι τεχνικά θέματα, αλλά και εξόχως πολιτικά. Το που δηλαδή πάνε τα λεφτά σου. Ναι. Συγκεκριμένα, να επανέλθω στο άρθρο 265. σε σχέση με το 125. Μεταφορά πόρων σε μέσα τα οποία θεσπίζονται υπό αυτόν τον κανονισμό για συγκεκριμένους τομεακούς κανονισμούς. Αυτό το άρθρο πιστεύουμε ότι πρέπει απλούστατα να διαγραφεί, γιατί αυτή η έννοια της μεταφοράς κονδυλίων είναι εκτός θέματος. Δεν είναι βεληξία, δεν είναι απλούστευση αυτό το πράγμα. Και μιλάει για μεταφορά κοντιλίων από στόχους ε, και προγράμματα για τα νέα καταπιστεύματα, για τα νέα ταμεία. Και αυτό μπορεί να γίνει και με τους κανονισμούς που προβλέπονται στις, στη συγκεκριμένη παράγραφο. Αυτό συνδέεται και με το άρθρο 38, που είναι καινούριο άρθρο, που αφορά το τμήμα των διαθωτικών και επενδυτικών ταμείων, που κατέτησε το κρατών μελών και με συμφωνία της Κομισιόν μπορεί να μεταφερθούν σε ένα ή περισσότερα μέσα ε, που θεσπίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Και αυτό είναι το θέμα του κατά την απόψή μας, της υποτιθέμενης ευελιξίας και απλούστευσης. Για τα τέσσερα ταμεία, τα οποία είναι της άμεσης αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, να αναφέρω το Ταμείο Απασχόλησης και κοινωνική Ένταξης. Εδώ οι προτινόμενες τροπολογίες των δεικτικών ποσοστών για την ετήσια χρηματοδότηση τριών αξώνων του Ταμείου και η αφαίρεση των ποσοστών για τους συστηματικούς τομείς των διαφόρων αξώνων είναι εντελώς απαράδεκτο κατά την απόψή μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να απορριφθεί. Δεν δικαιολογείται, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο και περιορίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου θεσπίζοντας στη θέσπιση προτεραιοτήτων της Ένωσης ε, με τα προγράμματα αυτά. Κάτι που είναι εντελώ απαράδεκτο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πέρα από την ε, έλλειψη δικαιολόγηση για τι 13, των άρθρων 13 και 14, δεν ξέρουμε πώ η τροπολογία του παρατήματο 1 θα διευκολύνει την πρόσβαση για κάποιε ομάδε στόχου στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και έχουμε πρόβλημα για του τρει δείκτε, ε, το εξέφασαν και οι κοινωνικοί εταίροι. Παρ' όλα αυτά, εάν τροποποιηθούν, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά αν θα πρέπει να τους αλλάξουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει. Πάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Προβληματικό. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη διαγραφή του ισχύοντος μηχανισμού στο άρθρο 15.2 για την ε, διάσωση συμφωνιών ε, μέσω του τριλόγου ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Εδώ φύγονται τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Και το Ταμείο τώρα για τους πλέον ενδεείς, για τους απόρους. Πολλέ από τι προτάσει που υποτίθεται προωθούν την απλούστευση, ενδεχομένως την προωθούν, αλλά πρέπει να τις ξανασκεφτούμε. Παραδείγματος χάρη το 42.3 η φρασιολογία δημιουργεί πρόβλημα για τη σημασία της τροποποιημένης ε, ε, φρασιολογία και τις επιπτώσεις που θα έχει στου τομεακού κανονισμούς. Επομένως, Πρόεδρε, αυτές είναι οι βασικές μας σκέψεις, βασίζονται στις αρχές μας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για τις τροπολογίες. Ε, καταληκτικά θα, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε τεράστια θέματα για την ε, αποδοχή τέτοιων κατώνων. Πώς μπορείτε να κάνετε τέτοιες πολιτικές, μάλλον αλλαγές πολιτική και να τις μεταμφιέζετε ε, σε, με τεχνικούς κανόνες. Παρουσιάζεται για τεχνικούς κανόνες, αλλά δεν είναι. Είναι πολιτικές αλλαγές. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Κυρία Τρεβίσο δεν είναι εδώ. Ποιο την αντικαθιστά από το ECR, Ουδής. Ο κ. Σελίμοβιτς από τους φιλελεύθερους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις τροπολογίες και την έκθεση που θεωρώ ότι είναι σωστή στη βαστής. Υποστηρίζω τις φιλοδοξίες της Επιτροπής που θέλει να πετύχει περισσότερη ευελιξία και απλούστευση. Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά και ορθά αυτά τα ταμεία. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που αναφέρθηκε με τις μεταφορές ε, κονδυλίων αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εκτός ε, εφαρμογής, αλλά ότι απαντάει στο ερώτημα που θέλω να θίξω. Στο πρώτο της προηγούμενης περίοδου η αξιολόγηση καταδεικνύει κάποιες προτεραιότητες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια μετανάστευση, προσφυγή κρίση, έκτακτες περιπτώσεις, ε, θέματα εσωτερικής ασφαλείας, η κρίση στην ε, γεωργία, το ψηλό επίπεδο ανεργίας, ε, κυρίως στους νέους και θεωρώ ότι θα πρέπει να ανασχεδιάσουμε τις προτεραιότητες αυτών των ταμείων. Οι δυνατότητες μεταφοράς είναι μία δυνατότητα που μας δίνει την ευκαιρία να πετύχουμε καλύτερα τον ασχετισμό των προτεραιοτήτων ε, σύμφωνα με την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι κακό. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Κάποιος να λαμβάνει κάποιο ποσό θα πρέπει τα μισά να τα δίνει σε κάποιον άλλον που θα τον βοηθήσει να ε, εκπληρώσει τις ε, διοικητικές του υποχρεώσεις. Και εφόσον αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση, θεωρώ ε, ότι πρέπει να εξέλθουμε από αυτήν. Πριν από μερικούς μήνες ε, αναφέραμε όλες τις διοικητικές υποχρεώσεις που πρέπει ε, κάποιος να εκπληρώσει για να λάβει το κονδύλιο. Ε, έγινε μία έκθεση σχετικά με αυτό και ήταν πραγματικά εργοτέχνης αυτή η έκθεση. Επομένως, συμφωνώ πλήρως με την ιδέα της απλούστευσης των μεθόδων και των κανόνων σχετικά με τα μία. Τέλος. Και όσον αφορά το τομέα για την παγκοσμιοποίηση, υποστηρίζω τους εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτία ε, των προβλημάτων που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Από ποια πολιτική ομάδα και αν προερχόμαστε, γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, τότε δίνουμε έδαφο στου λαϊκιστέ που τα εκμεταλλεύονται. Έχω δει την χρήση των ταμείων αυτών ad hoc κατά τη διάρκεια της θητείας μου, τρέχοντας από το ένα σημείο στο άλλο, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση και να ανταγωνιζόμαστε παράλληλα με τις τραγωδίες ε, που έχουν συμβεί. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά, και να εξοπλίσουμε σύμφωνα με αυτό τα ταμεία αυτά και σύμφωνα με αυτά που αναμένουμε να προκύψουν εξαιτία τη παγκοσμιοποίηση. Και επίσης να αναλογιστούμε ποιε είναι οι προτεραιότητες και να ζητήσουμε την αναθεώρηση των ταμείων και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Πιμέντα Λόπες, ο Ζώο απουσιάζει. Και η Μόνικα Βάνα. Από την FTD, κανείς. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντομινίκ Μαχτά. Ευχαριστώ. Ένας λαϊκιστής θα μιλήσει τώρα για να απαντήσει στον αγαπητό μας συνάδελφο που θεωρεί ότι όταν απαντάει στις ερωτήσεις απαντάει στους λαϊκιστές. Θα έρθει η μέρα που θα καταλάβετε ότι εσείς φταίτε για όλα αυτά αγαπητέ ε, κύριε και ότι συνενείτε με όλα αυτά. Ε, κύριε Σιγητά, αγαπητέ κύριε Λαβρίγε, Λαβριέ, Α, όχι, ο Λαβριέ κάτι αυτοκίνητα έφτιαχνε, εσείς κάτι σκάνδαλα κουβαλάτε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Λαβρίου, σας παρακαλώ να προεδρεύσετε. Εδώ είναι κοινοβούλιο. Πρόεδρε, να, να μην μου κόβει συστηματικά το λόγο ο κύριος Λαβρίου. Κύριε Μαχτά, σας παρακαλώ να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Μπορούν να σταματήσουν να μου κόβουν το λόγο κάθε φορά που μιλάω. Δεν σας κόβω κανένα λόγο, μιλάω στην πρόεδρο. Ωραία, και εσεί μιλάτε στου βουλευτέ. Όταν μιλάτε σε βουλευτέ, μιλάτε δια της Προέδρου σε μια επιτροπή. Παρακαλείται ο κύριο Μαχτά να επικεντρωθεί στην έκθεση που μα αφορά, ε, αντί να κάνει αυτά που έκανε σε προηγούμενη συνεδρία σε εις βάρος σα. Εγώ θέλω να τον καλέσω στην τάξη, ε, Εκείνο μου κόπτει το λόγο, με διακόπτη. Ζήτησα το λόγο, δεν σα έδωσε κανεί το λόγο. Λοιπόν, κύριε Ντομινίκ Μαρτά. Ναι. Εάν ένα μέλος κοινοβουλίου χρησιμοποιεί τη λέξη λαϊκιστής, αυτό αξιολογείται από τον καθένα μας ξεχωριστά και θα πρέπει ο καθένας να και αναλογιστεί. Είμαι λαϊκιστής. Εσείς θυμούσατε επειδή σας είπα λαϊκιστή. Φτάνει κυρία Πρόεδρε. Κάθε φορά μεροληπτείτε κυρία Πρόεδρε. Κάθε φορά μεροληπτείτε. Μόνο εμένα να καλείτε στην τάξη. Εγώ θα σας ζητήσω να αποχωρήσετε. Με αποκάλεσε λαϊκιστή και απαντώ. Ε, κάνω λάθος το όνομά του και ε, με διακόπτει. Κυρία Πρόεδρε, αυτά είναι συστηματικά. Έτσι γίνονται τώρα. Λοιπόν, δύο τεινά έχουμε τώρα. Είτε θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση με ησυχία και τάξη, είτε θα αποχωρήσετε τις αιθούσεις αν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε. Τι να σεβαστώ. Αυτός ο κύριος εδώ με διακόπτει. Εκείνος με διέκοψε και έχουν γράψει και οι κάμερες ότι με διέκοψε εκείνος εκείνος μπορεί να με διακόπτει. Ναι, αλλά μιλούσε και το διακόψατε κι εσείς και εκείνος έχει το δικαίωμα. Όταν μίλησε ο εισηγητή, δεν τον διέκοψα. Με αεροληπτείτε πρόεδρε κάθε φορά. Όχι, δεν πάω πουθενά. Εκείνος με διέκοψε. Ωραία, αναφέρεται να με, να με ε, απομακρύνουν δια της βίας. Τραβάνε και κάμερες, θα σπάσουμε και πλάκα. Απίστευτα αυτά, δεν το λέτε και συζήτηση κοινοβουλευτική. Κύριε Σαγητά, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να συνεχίσετε. Ε, κυρία Πρόεδρε, με, όση ώρα θέλετε. Καλά, δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω. Θέλω να απαντήσω στα σχόλια του κυρίου Πυρίνσκη, ο οποίος χρειάστηκε να βγει. Θα το δω διμερώς μαζί του, λοιπόν. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στο επεισόδιο που ζήσαμε εδώ και που είναι διαρκές. Ε, εγώ απλώς είπα στον κύριο Μαρτά, που ξέρει απολύτως πώς προφέρεται το όνομά μου, γιατί είπε ότι έχουμε κάμερες και δεν υπάρχει και πρόβλημα ε, μετάφρασης. Δεν λέγομαι λαβριέ, λέγομαι λαβριού. Και ήθιστε να μην κατακρεοργούμε τα ονόματα κανενός. Δεν θα τον έλεγα εγώ ποτέ διαφορετικά τον κύριο Μαρτά δεν το ε, επετέθην. Λυπάμαι για τον τόνο και το ύφο που πήρε η συζήτηση. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τι έχει να πει επί της ουσίας ο κύριος ε, Μαρτάν, που σίγουρα έχει τη βάση και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλου του βουλευτέ. για να δούμε εάν συμφωνούμε για κάποια πράγματα και διαφωνούμε σε κάποια άλλα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εις εξέταση αυτού του κειμένου πέρα από αυτά τα δικολαβικά που μπορούν να τα κάνουν στην Ολομέλεια γιατί φαίνεται είναι πολύ ενδιαφέρον που έχει κάμερες και στην ε, Ολομέλεια μπορεί να έχει και περισσότερους θεατές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι χώρος εργασίας και εργαζόμαστε ε, σε βάθος. Αν θέλει ο κύριος Μαρτέ να έρθει να με δει να συζητήσουμε την ουσία των θεμάτων και τις προτάσεις άκρος επικοδομητικές και ενδιαφέρουσες που έχει να κάνει, να το πράξει. Και δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, αν συμφωνούσαμε σε όλα θα ήμασταν στην ίδια πολιτική ομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς, αν θέλει, ε, όταν θα καταλαγιάσω λίγο τα πνεύματα, είμαι στη διάθεσή του, όπως και στη διάθεση όλων των άλλων ε, συναδέλφων βουλευτών. to... Ε, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία Γκρισάρ, αν δεν απατώμε, παρακαλώ. Φτάνει κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος εδώ, για να ακούσει τη διερμηνία, επειδή συμφώνησε μια συνάδελφος, πιο σόκαρε αυτό, δεν ήταν ούτε επιθετικό ούτε τίποτα, τι λέει ο κύριος, επειδή ε, συμφωνεί η συνάδελφός μου, την υβρίζει ε, λέγοντας να ποιοι είναι οι φίλοι και να ποιοι είναι οι πονηροί. Ε, τώρα αυτό τι είναι, σχολείο, δημοτικό ή κοινοβούλιο aura vu que c'est moi qui provoque dans cette salle. Όλοι κατάλαβαν ότι εγώ προβοκάρω εδώ πέρα. Καλά, άσε τώρα. Τι να συζητήσουμε τώρα, απόγευμα, ίσως άλλη μέρα είμαστε καλύτεροι. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλια. Ε, Κατακράσαμε τα σχόλια και περιμένουμε τις τροπολογίες με ανυπομονησία. Ευχαριστώ. Στάινρουκ. Στάινρουκ. Επειδή δεν ήμουν παρούσα την τελευταία περίοδο, ήμουν ε, εισήτρια για το πρόγραμμα EASY και η εντύπωση μου είναι ότι δεν έχει να κάνει με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αλλά με το γεγονός ότι η Επιτροπή της μη τροπολογίες προσπαθεί να αλλάξει από την πίσω πόρτα. Αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο με αποφασιστικότητα άλλαξε την πρόταση της Επιτροπής. Στο σχέδιο τα ποσοστά για το progress, τα ποσοστά δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κοινωνική ένταξη και εργασιακές συνθήκες, μικροχρηματοδότηση και μικροπιστώσεις και το ΟΕΡΕΣ, προγράμματα κινητικότητας και υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα ορίσαμε όλα αυτά. Και τώρα θέλει μέσα από αυτήν την πρόταση η Επιτροπή να πάμε στην αρχική πρόταση που είχε κάνει αυτή, και που αλλάχθηκαν ε, στον ε, τρίλογο με το Κοινοβούλιο. Αυτό ε, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις αυτού του Κοινοβουλίου δεν πρέπει εκ των υστέρων καθυστερημένα να επαναπροωθούνται στην Επιτροπή. Η συνάδελφος εργάζεται και αυτή εκεί επειδή δεν υπήρξαν προπτικές για το μέλλον ε, στα άλλα τα προγράμματα, το συζητήσαμε αυτό και θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα στο μέλλον πώς μπορούμε από κοινού ως κοινοβούλιο, όπως το κάναμε με το EASY, την πρόταση της Επιτροπής και αυτό που θέλει να ξαναπετύχει, όπως το αλλάξαμε τότε, να μπορέσουμε και τώρα να το στήριξουμε γιατί αυτό αφορά τα σημεία των προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση ε, ατόμων από τρίτες χώρες στην αγορά εργασίας. Είναι θέματα στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Πρόκειται για άλλα προγράμματα και γι' αυτό παρακαλώ τους συναδελφούς να δούνε ποια είναι η πραγματική πρόθεση της Επιτροπής πίσω από όλο αυτό. προσπαθεί να μας επιστρέψουν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και να θέσουν σε κίνδυνο την ε, διασυνορική συνεργασία. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαφριέ, δεν θέλω. Δεν έχω να πω τίποτα θα συναντηθούμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό και να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στις διάφορες απόψεις. Ε, ε, προθεσμία για τις τροπολογίες 28 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, οθέτηση στην ε, Επιτροπή Επασχόλησης, 2 και 3 Μαΐου, στις 11 Μαΐου στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή και η στην Ολομέλεια μετά το καλοκαίρι, στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου του 17. Τώρα. Έχουμε μια συνάντηση στη 4B 001. Είναι μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα συνεδριάσουμε στην αίθουσα της Επιτροπής, συγγνώμη, νομικών υποθέσεων για την ε, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις και θα συζητήσουμε επίσης και το καθεστώς για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην αλληλεγγύη με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτό θα γίνει στις 5 η ώρα αυτή η κοινή ακρόαση. Να πάτε εκεί, γιατί τα μέλη της Επιτροπής μας μπορούν να λάβουν το λόγο σε αυτήν την ακρόαση. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε πάλι με μία ε, συνάντηση σε μία άλλη αυσό, στη δική μας. Θα κάνουμε μια κοινή συνάντηση για τα προσόντα με την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, την Επιτροπή Πολιτισμού, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν πώς μεταχειριζόμαστε με τους δε όταν μας φέρνει ο κόσμος εδώ στο Κοινοβούλιο.